Okay, colleagues, if people can now... Καλώς συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Θα πάμε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης, ανταλλαγή απόψεων για την ε, πρόοδο με, σχετικά το, με τους ε, στόχους αηφόρου ανάπτυξης και τους δείκτες για αυτούς. Για τους δείκτες θα μιλήσουμε σήμερα. Για τους δείκτες των στόχων Sustainable Development Goals. Όταν ε, ήμασταν στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχαμε τη χαρά και την τιμή να συναντήσουμε τον Τζον Πούλιντζερ. Ε, συνάδελφοι, εσείς εκεί πίσω ε, που συσκέπτεστε, παρακαλώ να το κάνετε εκτός εθούσης ή να μιλήσετε πιο χαμηλόφωνα για να μπορούμε να ακούμε τους ομιλητές μας και να έχουμε σωστές ε, συζητήσεις. Ο κύριος Τζον Πούλιντζερ λοιπόν είναι επικεφαλής της στατιστικής υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι εθνικός στατιστικολόγος, προείδρευσε στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο ήταν επικεφαλής ε, όλης αυτής της ομάδας που κατάρτισε τους δείκτες. Εύκολη ήταν η υιοθέτηση των 17 στόχων, όλοι όμως οι υποστόχοι θα πρέπει να ε, επιτευχθούν και για να ε, τους επιτύχουμε πρέπει να είμαστε σε θέση να ξέρουμε πώς θα τους μετρήσουμε. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερος που είναι εδώ και είναι, συνοδεύεται από την ε, Μπάρμπαρα Πέσε Μοντέρο, διευθύντρια του γραφείου UNDP στις Βρυξέλλες. Θα ξεκινήσουμε με μια παρουσίαση του κυρίου Πούλιντζερ, της δουλειάς που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Θα μας μιλήσει για τους δείκτες, για τα διάφορα θέματα που άπτονται αυτών και ελπίζουμε να ακούσουμε ε, από τον κύριο Πούλιντζερ και ε, κάτι για τα επόμενα βήματα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που είμαι στην Επιτροπή εδώ σήμερα. Επιτρέψτε μου όμως να ξεκινήσω με τη συνεδρίαση της Νέας Υόρκης και να σας πω ότι πριν από τη Γενική Συνέλευση το Σαββατοκύριακο προηγήθηκε, συναντήθηκα με την Επιτροπή Και ήταν πραγματικά εξαιρετικές οι ημέρες αυτές. Όποιος ήταν παρόν από εσάς τότε ε, σίγουρα το ένιωσε. Και τα δύο πιο χαρακτηριστικά ε, θέματα του Σεπτεμβρίου, τα οποία σχετίζονται με τη συζήτηση μας σήμερα, ήταν τα εξής. Πρώτον, το εύρος της πολιτικής βούλησης και φιλοδοξίας, έτσι ώστε κανείς να μην υστερήσει, κανείς να μην μείνει πίσω. Και δεύτερο, κάτι που μας αφορά ιδιαίτερος, είναι το πόσο επικρατούσε η ιδέα ότι είμαστε στην έναρξη μιας ε, επανάστασης σε σχέση με τα δεδομένα. Και αν καταφέρουμε να αντιθασσεύσουμε αυτή την εξέλιξη, θα μπορέσει ο κόσμος να πάρει καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον. Ναι, εγώ μίλησα ως πρόεδρος της Επιτροπής αυτής της στατιστικής. Ζήτησε ο πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης να συγκροτηθεί η Επιτροπή και να έχουμε δείκτες για κάθε στόχο και για κάθε υποστόχο. Ο συνάδελφος από τη Βρασιλία έχει αναλάβει τα ενιαία της Επιτροπής και εγώ τώρα είμαι αντιπρόεδρος αυτής. Το Μάρτιο του 2015 συνήλθε η Συστατιστική επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών και εξέτασε αυτό το θέμα των δικτών και δύο είναι τα πεδία εργασίας. Πρώτον, να ανταποκριθούμε στην τεχνική πρόκληση να δώσουμε ορισμό για τους δίκτες και δεύτερον, να εξετάσουμε το θέμα του capacity building. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ενδιαφέρεται για αυτή, γι' αυτό θα μιλήσω καταρχάς για τους δείκτες. Στη συνεδρίαση του Μαρτίου 2015, η Στατιστική Επιτροπή των Εθνών δημιούργησε μια υπηρεσία και μια ομάδα εμπειρογνωμόνων με συμπροέδρου του συναδέλφου από Μεξικό και Φιλιππίνε. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων έχει κάνει εξαιρετική δουλειά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα έχει εμπλέξει εκπροσωπούς πολλών χωρών λειτουργεί με διαφάνεια, συμπεριλαμβάνει τους πάντες, κάνει διάφορους γύρους διαβουλεύσεων και παρουσίασε μια δέσμη 131 δικτών στην Επιτροπή των Εθνών που συναντήθηκε το Μάρτιο φέτος και αυτό είναι το σημείο έναρξη, σημείο κίνησης για να προοδεύσουμε και να προχωρήσουμε ακόμα πιο πέρα μαζί με το υπόλοιπο πρόγραμμα εργασιών τη της ομάδας των εμπειρογνωμόνων. Έχει μπει αυτή η δέσμη μέτρων στην ε, αλυσίδα εξέταση και ακολουθεί τη διαδικασία στους κόλπους του ΟΗΕ και θα φτάσει να εξεταστεί και σε πολύ ψηλό επίπεδο βεβαίως. Τώρα, θα κατηγοριοποιήσουμε τους δείκτες αναλόγως με το πόση δουλειά χρειάζεται ο καθένας για να αναπτυχθεί πλήρως και κατά πόσο ταιριάζει για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχουν υφιστάμενοι ορισμοί έτοιμοι, υπάρχουν έτοιμα διαθέσιμα δεδομένα. Και γι' αυτό η ομάδα περιγνωμών έχει συστήσει υποομάδες. Μία για την αποσύνδεση των δεδομένων, τον καταμερισμό τους, αυτό ενδιαφέρει τη δική σας επιτροπή, την ανάλυση δηλαδή αυτών και αν ε, π.χ. με κριτήρια εσόδων, φύλου, μεταναστευτικού καθεστώτος, γεωγραφικής τοποθεσίας, ε, ηλικίας, εισοδήματος, ε, μεταξύ άλλων. Δηλαδή υπάρχει ένα πολύ ισχυρό αίτημα για δεδομένα, ε, όπως φαίνεται. Άλλη υποδομάδα της ομάδας υπερηγνωμόνων κοιτάζει τις διασυνδέσεις. Μπορεί, για παράδειγμα, μια ομάδα δικτών να μας βοηθήσει να πετύχουμε περισσότερους από έναν στόχους, π.χ. δημογραφικοί δείκτες. Μία άλλη ομάδα ασχολείται με τη μετάδοση των δεδομένων. Έχει αναπτύξει έναν μηχανισμό, τον SDMX, που έχει εφαρμοστεί ευεραίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχει και πιο ευρείες εφαρμογές και ε, βοηθάει έτσι ώστε να συγκεντρωθούν τα διάφορα δεδομένα που χρειάζονται για να μπορεί να γίνει reporting, ε, αναφορά και έκθεση σε επίπεδο εθνικό, διαπεριφερειακό, περιφερειακό, τοπικό, διεθνές κτλ. Πολύ σημαντικό είναι να δούμε και τη διασύνδεση μεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών επιπέδων. Θα έπρεπε λοιπόν και έπρεπε χρειάστηκε να ε, βάλουμε στο ίδιο καλάθι τη δουλειά των κρατών μελών, ε, άλλων ειδικών φορέων όπως είναι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η Παγκόσμια Τράπεζα ή ε, ε, το UNDP, να βάλουμε στο ίδιο καλά την ίδια τη δουλειά του ΟΗΕ, αλλά και το έργο που έχει παραχθεί στα πανεπιστήμια, στην οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, στα διάφορα ερευνητικά Ινστιτούτα απανταχού στον κόσμο. Το σημαντικό είναι να μην χάνουμε το σημείο εστίασης και να έχουμε ένα κοινό πρόγραμμα. Θα συνεχίσουμε την, να κατευθύνουμε αυτή την εργασία και θα υπάρξει ένα πρόγραμμα εργασιών που θα δημοσιευθεί επισήμως το Μάρτιο του 2017 από την ομάδα εμπειρογνωμόνων. Μέσα σε αυτό το πνεύμα των στόχων ε, για την αηφόρο ανάπτυξη και κυρίως το στόχο 17 είναι η ανάγκη να υπάρξουν επενδύσεις για την υλοποίηση αυτών των στόχων, δηλαδή χρηματοδότηση για ανάπτυξη. Και αυτό τονίζει το πόσο σημαντικό είναι να αναλύουμε τα δεδομένα με κριτήρια υψηλής ποιότητας. Δίδεται προτεραιότητα στο capacity building στις ε, ε, μικρές νησιωτικές χώρες κυρίως, αλλά και στις χώρες που είναι αποκλεισμένες από τις θαλάσσιες οδούς, μεταξύ άλλων. Στη Νέα Υόρκη ασχολήθηκαν ιδιαίτερος πρόσφατα με το θέμα του capacity building για δεδομένα. Και το βασικό ζήτημα πάνω στο τραπέζι ήταν το κενό ανάμεσα στους 231 δείκτες που στηρίζει το NSC και ε, το, τη δουλειά που χρειάζεται από πλευράς χρηματοδότησης αλλά και στην πράξη στις διάφορες χώρες. Η Επιτροπή λοιπόν τον Μάρτιο του 2015 συγκρότησε μια ομάδα εμπειρογνωμένων με προέδρους από την Ακτήση Ελεφαντοστού και την Ουγγαρία με σκοπό να εξετάσουν το συντονισμό, της εταιρικέ σχέσεις και το capacity building όλων αυτών μετά το 2015 για να υπάρχει σωστή συνέχεια και παρακολούθηση και κατέληξαν σε συμπεράσματα. Πρώτον, Πρέπει να επενδύσουμε στα εθνικά στατιστικά συστήματα. Αυτό ήταν βασικό συμπέρασμα, γιατί τα εθνικά στατιστικά συστήματα δεν συνεχίζουν να προσφέρουν επαρκή δεδομένα και πρέπει να στηριχθούν για να γίνουν μέλη μιας κοινότητας δεδομένων και τελικά αυτή η κοινότητα δεδομένων θα είναι και ο καταλήτης για την έλευση των αλλαγών. Οι παραδοσιακές πηγές λοιπόν των επισήμων δεδομένων σίγουρα χρειάζονται και θα συνεχίσουν να χρειάζονται και υπάρχουν όμως και νέες πηγές δεδομένων που είναι και αυτές χρήσιμες. Ο συνδυασμός είναι το πιο σκόπιμο, ο πιο σκόπιμος ε, εύλογος τρόπος δράσης έτσι ώστε να υπάρξει κοινότητα δεδομένων και να ενισχυθεί ε, η επιστημονική τεκμηρίωση όλων αυτών. Χρειάζεται οι κυβερνήσεις να έχουν τη δυνατότητα να αναλύουν τα δεδομένα. Γιατί είναι βασικός πόρος για τις κυβερνήσεις τα δεδομένα, ώστε να πετύχουν τους στόχους τους και κυρίως τους στόχους της ατζέντα για το 2030. Για να είμαστε αποτελεσματικοί πρέπει να, έχουμε, ε, να αυξήσουμε τη ζήτηση ε, των πελατών, των χρηστών για τα δεδομένα αυτά. Και θα πρέπει σε αυτό το εγχείρημα να εμπλακεί και ο ιδιωτικό τομέα και η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Να έχουμε ευρύ πνεύμα, ανοιχτό, να έχουμε πρωτοβουλίε ε, και να δούμε ποια έχει τι περισσότερε πιθανότητε να πετύχει σε συνέργεια με Ινστιτούτα και ερευνητικά ιδρύματα. Η ελοχεύει ο κίνδυνος οι λίγοι πόροι να μην χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά και η προσπάθεια τελικά να κατακαιρματιστεί και να χάσουμε από, την, ε, ε, από τα μάτια μας το στόχο. Θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Τέλος, η ανάπτυξη δεξιοτήτων θα είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό και η ικανότητα μετάδοσης της γνώσης. Τα σκληρά, δύσκολα προβλήματα μπορούν να λυθούν μόνο ε, μία φορά δεν χρειάζεται να ξαναπροκύψουν όταν και εφόσον διαδίδεται η γνώση. Στόχος είναι να έχουμε βιώσιμες δυνατότητες που θα ε, διαρκούν σε βάθος χρόνου σε όλα τα έθνη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε ένα data campus. Ορίζουμε και συνδέουμε τα διάφορα ιδρύματα και τα συστήματα μεταξύ τους και στηρίζουμε τα συμπεράσματά τους. Είναι εξαιρετικά τεχνική η παρακολούθηση αυτή της εξέλιξης, αλλά ελπίζω να είναι χρήσιμη στην Επιτροπή σας. Ευχαρίστω θα δεχτώ τις ερωτήσεις σας και θα ακούσω τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ, Τζον. Θα δώσω το λόγο αμέσω ε, στον συνάδελφο να μας πει τι θα γίνει από πλευράς πολιτικής, ε, ποια είναι τα επόμενα βήματα σε ό,τι αφορά τους βιώσιμους στόχους, ε, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για να έχουμε μια πλήρη εικόνα και να δούμε πώς μπορούμε να επηρεάσουμε. Η Μπάρμπαρα. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που επανέρχομαι εδώ στο Κοινοβούλιο. για να συνεχίσουμε ε, το διάλογο, γιατί από κοινού παρακολουθούμε την κατάσταση και θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να επηρεάσουμε και να συμβάλλουμε σε αυτή την όλη συζήτηση. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά που ήρθα, ο στόχος μας πέρυσι ήταν να πετύχουμε τους στόχους και νομίζω ότι καθοδηγήσαμε την όλη διαδικασία με επιτυχία ως Ευρώπη. Τώρα έχουμε μπροστά μας την εφαρμογή. Υπάρχουν διάφορες συμφωνίες όπως ε, για τις στατιστικές, για παράδειγμα, που ισχύουν και φέτος. Αυτό που θέλουμε είναι να μην χάσουμε την ορμή και η ενέργεια, η θετική ενέργεια που κινητοποιήθηκε πέρυσι θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει και ήδη ξεκινάμε να βλέπουμε αποτελέσματα επιτόπου. Και πράγματι Πολύ θετικά βλέπουμε το γεγονός ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ε, βλέπουν ε, και ε, πανεξετάζουν τι σημαίνει όλο αυτό. Βέβαια υπήρχαν δύο-τρεις μεγάλες διαφορές με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης σε σχέση με τους προηγούμενους. Και η πρώτη διαφορά είναι ότι είναι οικουμενική η στόχη και σίγουρα αυτό επηρεάζει γιατί όλες οι χώρες ήθελαν να συμμετάσχουν και όχι μόνο ευρωπαϊκές και βέβαια θέλουμε να έχουμε συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία που θα μπορούν να ανταλλάσσουν οι χώρες ε, ανεξαρτήτως επίπεδο ανάπτυξης ή υπήρου στην οποία ανήκουν. ανάπτυξη ή η στόχη. Άρα, κανείς δεν θέλουμε να μείνει πίσω και αν δεν θέλουμε να μείνει κανείς πίσω, θα πρέπει και αυτοί να υπάρχουν, να φαίνονται και να μετρηθούν να ληφθούν υπόψη σας τα εθνικά στατιστικά στοιχεία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για κάτι που πρόσφατα συζήτησα, ε, χάρη για την κοινότητα των Ρωμά στην Ευρώπη, που φαίνεται σε πολλά εθνικά στατιστικά στοιχεία να μην υπάρχει καν και σίγουρα ε, είναι μια κοινότητα που κανείς δεν θέλει να τους αφήσει εκτός στην Ευρώπη. Και υπάρχουν και άλλες τέτοιες ομάδες. Θέλουμε λοιπόν να συμμετέχουν στις πολιτικές, ε, να είναι τμήμα των πολιτικών και έτσι όπως εξελίσσεται η πολιτική πρέπει να περιλαμβάνονται αυτές οι ομάδες και το πρώτο βήμα είναι τα στατιστικά στοιχεία για να δούμε ποια είναι η γραμμή αφετηρίας, η baseline όπως λέμε στα στατιστικά και μετά να δούμε τι πολιτικές εφαρμόζονται και ποια είναι τα επίπεδα, το βιωτικό επίπεδο κτλ. Είναι σημαντική αυτή η χρονική στιγμή στην οποία βρισκόμαστε, διότι συνεχίζουμε ουσιαστικά να δημιουργούμε το πλαίσιο και όπως είπα πολύ σημαντικό είναι και το στατιστικό πλαίσιο, αλλά είναι σημαντική η στιγμή αυτή η χρονική γιατί τον Ιούλιο έχουμε και τα βήματα συζήτησης, ε, το φόρουμ που θα αρχίσει να συζητεί αυτό το θέμα. Τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες εθελοντικά θα παρουσιάσουν τις εκθέσεις τους, ε, μία είναι η Γερμανία, άλλη είναι η Γαλλία, και οι άλλες δύο είναι η Φινλανδία και η Εστονία νομίζω. 20 χώρες θα παρουσιάσουν τελικά τις εκθέσεις τους. Είναι προκαταρκτικές βέβαια αυτές οι εκθέσεις. Γιατί θα δείτε και εσείς ότι μόλις συμφωνήθηκε το πλαίσιο, το στατιστικό και οι χώρες ξεκινούν να προβλημα... τον προβληματισμό για το πώς θα προχωρήσουν. Είναι σημαντικό όμως για εμάς αυτό το στάδιο, διότι θα δώσει καλά παραδείγματα και καλά παραδείγματα για το τι γίνεται και για το ποια είναι η πολιτική δέσμευση των χωρών. θέλουν να συμμετέχουν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το ότι η Γαλλία, η Γερμανία συμμετέχουν και δείχνουν τελικά ότι είναι σημαντική αυτή, αυτό το θεματολόγιο, αυτή η στόχη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό είναι σημαντικό και πω κάτι παρενθετικά. Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω και σας να ενθαρρύνετε τις κυβερνήσεις σας να συμμετάσχουν ε, στο φόρουμ σε υπουργικό επίπεδο, γιατί υπάρχει το τεχνικό σκέλος και μετά έχουμε και τριήμερο φόρουμ σε υπουργικό επίπεδο. Φοβούμαι ότι στην Ευρώπη πολλές φορές υπάρχει εντύπωση ότι το θεματολόγιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης δεν ε, αφορά και τόσο πολύ την Ευρώπη ότι πιο πολύ έχει να κάνει με τις όμενες χώρες. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Γιατί και το θεματολόγιο του 2030 και η αναπτύξη τη αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και κατανάλωση, την ενέργεια, την ένταξη, την φτώχεια, την απασχόληση κτλ. Όλα αυτά τα θέματα έχουν σημασία για την Ευρώπη ή οι διαφορέ των δύο φύλων. Μιλήσαμε για την απομαδοποίηση. Ε, θα δούμε όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν και τα στατιστικά και η Ευρώπη θέλει να αποδείξει ότι ηγείται σε πολλά μέτωπα και μπορεί να δίνει το καλό παράδειγμα. Ή σε άλλα ε, παιδιά θα πρέπει να δει η Ευρώπη τι προκλήσεις έχει να αντιμετωπίσει και πώς μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίε και δράσει όλου αυτού του τομεί. Άρα, επαναλαμβάνω, αυτό το φόρουμ είναι μια πολύ σημαντική χρονική στιγμή. Βέβαια, οι προσδοκίες είναι και στο του δυνατό επίπεδο για το φόρμα, εφόσον όπω είπα μόλι ξεκινούμε με αυτή τη διαδικασία, είναι μια πρώτη φάση για να δούμε πώς εκπονηθούν οι εκθέσει. Τα στατιστικά ακόμα είναι, θα έλεγα σε μεγάλο βαθμό, πειραματικά, αλλά αυτό είναι καλό ε, γιατί θέλουμε να δούμε ε, πώς θα το εφαρμόσουμε στην πράξη και τι μαθήματα μπορούμε να δώσουμε μετά και στους επόμενους, γιατί ο στόχο είναι να δούμε και οι χώρε τι έχουν και τι χρειάζεται ακόμη να αναπτύξουν για να μπορούν να υπονοούν τέτοιου είδους εκθέσεις. Εφτά είναι οι χώρε που έχουν ήδη ξεκινήσει και πολλέ ε, αναπτυσσόμενε χώρε. θα ήθελα να σα πω ότι είναι παράδειγμα για τι αναπτυγμένε χώρε που ακόμη δεν έχουν προχωρήσει στην πράξη. Αλγερία, Εκουαδόρ, Κολομβία, Ονδούρα, το Λάο, Μογγολία ήδη εξετάζουν τι στατιστικέ του βάσει για να δουν τι έχουν και αυτά τα στοιχεία που έχουν σε ποιο βαθμό είναι χρήσιμα και ποια στοιχεία ακόμη πρέπει να αναπτύξουν και ποια μπορούν να ανταλλάξουν με άλλες χώρες. Πριν από λίγο καιρό είχαμε πει ότι υπάρχουν κάποια συστήματα στην Λατινική Αμερική, στην Κολομβία για παράδειγμα, που θα μπορούσαν να είναι πολύ χρήσιμα για πολλές άλλες χώρες. Άρα η παρουσία σε αυτό το φόρουμ θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε αυτή τη συζήτηση και να είναι και σε πολύ επικοδομητική βάση. Επίσης είχαμε αναφέρει και τα Ηνωμένα Έθνη ως ένα χώρο συζήτησης όμως η ΟΗΕ είναι και ένας χώρος στο οποίο στηρίζουμε και πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Έχουμε το μηχανισμό MAPS, όπως λέγεται, που έχει να κάνει με τις εθνικές διαδικασίες, ε, τις στατιστικές, τα μεταξιακά προγράμματα, να λαμβάνεται η διάσταση και να δούμε πώς μπορούμε να επιταχύνουμε τα πράγματα. Η στατιστική είναι σημαντική και η πολιτική βέβαια είναι σημαντική και έχουμε και ένα πιλωτικό πρόγραμμα με 20 χώρες για να δούμε τι γίνεται σε αυτές τις χώρες και αν τις στηρίξουμε, αν θα προχωρήσει προς τα εμπρός τελικά πολύ πιο γρήγορα η ατζέντα των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε αυτόν τον διάλογο και με αυτέ τι χώρε και με την Κομισιόν, γιατί ελπίζουμε ότι πολλά από όσα διδαχθούμε θα μπορούσαμε να τα εντάξουμε στι δικέ μα πολιτικέ σε πολλά επίπεδα. Ξέρετε ότι έχουμε σύντομα, θα έχουμε σύντομα την ανακοίνωση. Άρα ο Ευρωπαϊκό Προβληματισμός θα ωφεληθεί τα μάλλον από, όλου αυτούς από όλα αυτά τα βήματα συζήτηση. Ω τελευταία παρατήρηση, να επαναλάβω κάτι που έχω ξαναπεί, αλλά θέλω να το επαναλάβω γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό. Διότι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης είναι πάρα πολύ σημαντική Βέβαια, απαιτούν μια διαφορετική εταιρική σχέση. Δεν θα περιουστούμε στις κυβερνήσεις. Ε, έχονται διάφοροι τομείς, κοινό των πολιτών, ο δυτικός τομέας, ε, τα μίντια, ε, αλλά και τα κοινοβούλια. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να είμαστε στο ίδιο επίπεδο, να είμαστε μαζί. Σίγουρα τα κράτη γκρίνουν τους προπολογισμού, θα παρακολουθούν και το τι γίνεται και είναι και καλύτερο ίσω χώρο συζήτηση και ανταλλαγή μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, τα κοινοβούλια. Παραλαμβάνω. Τον Ιούνιο έχουμε τα EDDs. Εκεί θα έχουμε την εξαρτία μας για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και εκεί θα δείτε πόσο σημαντικά είναι τα στατιστικά στοιχεία. Τα έχουμε δραστικές οθόνες με στοιχεία και με την πραγματικότητα. Γιατί τα στατιστικά δεν είναι αριθμοί. Μιλάμε για ανθρώπους, ε, ε, για γυναίκες, ε, για νέου. Ε, ηλικιωμένου, Εξετάζουμε τα οικονομικά μεγέθη και τις πραγματικότητες. Σίγουρα ε, πρέπει ε, να ληφθεί υπόψη και η τεχνολογία, αλλά εδώ μιλάμε για ανθρώπους, ε, για ανθρώπους με σάρκα και οστά και θα δούμε τα στατιστικά και στο πλαίσιο του ΙΕΓ, θα δούμε τους ανθρώπους, ε, τις πραγματικότητες, ε, τα νούμερα και θα το κάνουμε διαδραστικά. Γιατί το στατιστικό πλαίσιο για το μέλλον δεν ε, περιορίζεται σε νούμερα. Θέλουμε να είμαστε πιο καινοτόμοι στον τρόπο με τον οποίο συζητούμε για τους ανθρώπους, στον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε τις πληροφορίες και εκπονούμε στέρεα στατιστικά στοιχεία. Και κυρίως θέλουμε να έχουμε διαδραστικές μεθόδους και μπορούμε, υπάρχουν αυτές οι μέθοδοι σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ποιο συνάδελφο θέλει να πάρει το λόγο. Ελίσσες Λάιν και μετά η Μαρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και να ευχαριστήσω και τον κύριο Πούλινγκερ και την κυρία Πίσεμαν για την παρουσία τους εδώ σας καλωσορίζω κύριε Πουλιγκέρ. Συναντηθήκαμε στη Νέα Υόρκη ήδη μία φορά και πραγματικά είναι κρίσιμη σημασία η παρουσία σας εδώ, διότι θεωρούμε το ζήτημα αυτό μέγιστη σημασία. Εμείς σε αυτή την Επιτροπή πάντοτε τονίζαμε τη σημασία της πολύ ευαίσθητης δουλειά σας και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Όταν συναντηθήκαμε, μπορεί να θυμάστε ότι κάναμε τα δύσκολα ερωτήματα και εσείς κάνατε και θα ήθελα να συνεχίσουμε έτσι. Για μένα λοιπόν το ερώτημα έχει ως εξής. Ε, πόσο εύκολο ήταν να συνεχίσετε με τους δείκτες από τεχνική άποψη όταν γνωρίζουμε ότι υπάρχει και πολιτική, τόσο μεγάλη πολιτική σημασία αυτής της συζήτησης. Ε, πώς αυτό επηρέασε τη δουλειά σας μέχρι το τέλος. Αυτό με και στη δεύτερη ερώτησή μου. Μετά από εννέα μήνες ε, που πέρασαν από τότε που συναντηθήκαμε, ε, ποια είναι η γνώμη σας, ε, πώς ε, μπορέσατε σε τεχνικό επίπεδο να διαχειριστείτε αυτές τις πολιτικές συνιστώσεις και πόσο ε, ισχυρή είναι η θέληση να προχωρήσουμε βάσει αυτής της πολιτικής δέσμευσης και από το Ηνωμένα Έθνη από τη Γενική Συνέλευση. Μετά μιλήσατε για τα αναλυτικά στοιχεία. Γνωρίζουμε όλοι εδώ ότι όταν δεν μπορείς να μετρήσεις τα στοιχεία, στην ουσία είναι ανύπαρκτα, είναι αόρατα. Ειδικά όταν μιλάμε για θέματα φύλου, τα οποία όπως όλοι γνωρίζετε ε, είναι θέματα που επιδιώκουμε ιδιαίτερα να ρυθμίσουμε τώρα ε, και όταν μιλάμε και για ανισότητες. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε στοιχεία για αυτά. Το ερώτημά μου έχει ως εξής. Μας είπατε στη Νέα Υόρκη και εδώ πόσοι πολλοί συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, ε, μπήκανε ε, στη διαδικασία αυτή και με κυβερνητικές οργανώσεις και άλλοι κοινωνικοί οργανισμοί. Όμως ε, και στη συλλογή των δεδομένων καλό είναι να εμπλέκονται γιατί αν θέλουμε να κάνουμε όποια προσπάθεια απαιτείται για τη δημιουργία ικανοτήτων στις χώρες, διότι δεν υπάρχει αυτό το δυναμικό, αυτή η ικανότητα στις χώρες αυτή τη στιγμή, κάποιες χώρες μπορεί να ενδιαφέρονται να μάθουν πώς να συλλέγουν καλύτερα τα δεδομένα, γιατί όταν μαζέψεις τα δεδομένα, τότε βλέπεις τα προβλήματα. Τότε βλέπεις ότι δεν γίνονται αρκετές προσπάθειες όσον αφορά έναν στόχο ή τον άλλο. Ε, πόσο σημαντικό λοιπόν είναι να, εμπλακούν αυτές οι οργανώσεις στη συλλογή των δεδομένων. Ε, και κάτι τελευταίο, σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Μοντέρο. Ε, ζητάμε από την πρώτη μέρα να μας πείτε τι γίνεται με την εφαρμογή. Την ίδια ημέρα που εγκρίθηκε και αυτό το θέμα, αυτή η σε διάταξη στη Νέα Υόρκη, για την εφαρμογή των στόχων ε, συζητάμε αυτό. Δεν χρειάζεται το Ηνωμένα Έθνη να είναι απλώς ε, το 21ο ε, μέλος στα 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς στο Κοινοβούλιο θέλουμε να παίξουμε αυτό το δυνατό ρόλο, να προωθήσουμε την καθολικότητα που είναι το πιο σημαντικό στοιχείο αυτής της ατζέντα και την προσέγγιση αυτή που ε, ακολουθεί ε, αυτή η στρατηγική. Και επίσης να περάσουμε και πέρα από τις επιτροπές. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν είναι εδώ η Επιτροπή και θέλει να πει κάτι. Ίσως αργότερα θα, μπορέσατε να, θα μπορέσετε να μας δώσετε κάποια στοιχεία γι' αυτό. Γιατί στο τελευταίο Στρασβούργο Είχαμε τον Επίτροπο Τίμερμαρς που μιλούσε για τους στόχους και την ε, ολοκληρωμένη προσέγγιση. Οπότε ίσως η Κομισιόν θα μπορούσε να μας πει πράγματα και τα Ηνωμένα Έθνη θα μπορούσαν να μας να ακούσουν. Σας δίνω λοιπόν μια προειδοποίηση ότι θα μιλήσετε σε λίγο. Και η Μαρία Χόιμπουργκ. Ευχαριστώ ε, πολύ. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Μισό λεπτάκι, περιμένω να βάλετε τα ακουστικά σας. Ναι. Λοιπόν, περιμένω να μ' ακούσετε. Είπατε ε, ότι η Ευρώπη πρέπει να εφαρμόσει και πραγματικά θεωρώ ότι επιγόντως πρέπει να εφαρμόσει η Ευρώπη όχι μόνο στους τομείς ε, όπου ακόμα δεν είμαστε βιώσιμοι ή έχουμε ελλείμματα. Μυρίσαμε για το φύλλο. Υπάρχουν ε, τομείς στους οποίους υπάρχουν ελλείμματα, όμως στο μεταξύ υπάρχουν και δείκτες που δείχνουν ότι υπάρχουν και πολιτικές ε, διαστάσεις που ανέφερε και η συνάδελφος. Ε, σε ε, ζητήματα ας πούμε ε, που μπορεί να μην επηρεάζουν την βιωσιμότητα τη δική μας αλλά των άλλων. Θέλουμε λοιπόν δείκτες ε, ε, για να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις ε, αυτών που κάνει η Ευρώπη σε άλλες περιοχές του κόσμου. Αν επηρεάζει τη δική τους βιωσιμότητα, την εργασία τους και τους δικούς τους στόχους ανάπτυξης. Ευχαριστούμε την η Λόλα Σάντσες έχει το λόγο. Ευχαριστώ Λίνα. Πιο πολύ είναι σκέψη αυτό που θα πω. Έχοντας υπόψη την τρικουμενικότητα ε, του Ναθηματολογίου, όπως είπατε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να είναι υπόδειγμα στη διαδικασία. Να δείχνει δηλαδή πώς μπορεί να επιτευχθούν με συγκεκριμένους στόχους ε, ε, και αυτή, αυτά οι στόχοι. Αλλά δεν έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Ζητήσαμε συγκεκριμένη δράση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ψήφισμά μας και θεωρούμε ότι είναι Τέσσερα τα σημαντικά. Να υπάρχει πολιτική, ισχυρή πολιτική ηγεσία για να προωθήσει το θεματολόγιο, να είναι σαφή η στρατηγική εφαρμογή στη θεματολογία, να υπάρχουν επίσης επαρκή ε, οικονομικοί πόροι και σε ό,τι αφορά τη διαδικασία εφαρμογή, θα πρέπει να είναι συμμετοχική. Η κοινωνία των πολιτών, το είπε και η σύντροφο Σέλ, θα πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο. Είναι σημαντικό επίσης ε, να μην λησμονούμε άλλες αρχές ε, όταν ε, θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτούς τους στόχους, όπως είναι η αποτελεσματικότητα για τη βοήθεια επίσης, η παρακολούθηση ε, στις διάφορες χώρες, ε, η παρουσίαση, των δικτών για να μπορούν οι χώρες να ενισχύσουν τις εθνικές δομές και να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην όλη διαδικασία. Δηλαδή, να μην είναι μόνο οι διεθνείς οργανισμοί αυτοί που θα ελέγχουν και θα παρακολουθούν. Σίγουρα είναι σημαντικό το κόστος για όλα αυτά, εξού και χρειάζεται να, τεθούν, να διατεθούν όλοι όλοι οι απαραίτητοι πορεί, ιδίω για να φτάσουμε στο 0,7%. Και επίση θα πρέπει να κινητοποιηθούν περισσότερο οι εγχώροι πόροι. Η ερώτηση μου τώρα, η μόνη ερώτηση που έχω να αποβάλω είναι πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τις χώρες του Νότου να έχουν τα απαραίτητα μέσα και εργαλεία για να μπορούν να παρακολουθούν και να ελέγχουν από μόνα του τα κράτη. όπως είπα, όχι οι διεθνεί οργανισμοί μόνο να ελέγχουν, αλλά και τα κράτη-μέλη να μπορούν να ελέγχουν την υλοποίηση των στόχων. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θέλει κάποιο άλλο να έρθει στο λόγο, Κύριο Βέντα. Ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα στοιχεία που μας παρουσιάσατε σήμερα το πρωί. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ορισμένοι δείκτες για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίοι θα υποτίθεται ότι βασίζονται σε αξιόπιστα δεδομένα. Γνωρίζουμε ότι 72 από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ όμως δεν έχουν συμπηλήσει κανένα δεδομένο σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τη φτώχεια και αυτούς που ζουν κάτω από το κατόφλι της φτώχειας. Εδώ μιλώ κυρίως για χώρες που είναι σε πολύ ρευστή, σε πολύ ασταθή πολιτική κατάσταση από το παρόντο. Η ερώτηση μου είναι η εξή. Αν δεν έχουμε τέτοια δεδομένα, αν οι χώρε δεν διαβεβάζουν τέτοια δεδομένα, τι γίνεται. Είπατε χρήση, ε, συμπίληση δεδομένων κτλ. Αν δεν συνεργάζεται κάποιο, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Με ποιο τρόπο, αν υπάρχει, θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε την συλλογή δεδομένων και πώς θα μπορούσαμε να ε, επιβεβαιώσουμε την καταλληλότητα και την ακρίβεια των δεδομένων. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Νικολέτα Μελό, νομίζω, είναι εκπρόσωπος Κομισιόν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ που μας καλέσατε για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εμείς θεωρούμε ότι η υιοθέτηση της έκθεσης της Interagency και της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τους στόχους αηφόρου ανάπτυξης είναι κάτι το εξαιρετικό. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την υλοποίηση της ατζέντα, της πολιτικής ατζέντα για το 2030. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτά θα τα στηρίξει η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στο εγγύς μέλλον. Θεωρούμε ότι ο κατάλογος των μελλοντικών δικτών, παρόλο που επιδέχεται τελειοποιήσεων, αποτελεί μια πολύ καλή βάση εργασίας για να ξεκινήσουμε τη δουλειά και να προοδεύσουμε, να σημειώσουμε πρόοδο έναντι των ε, στόχων αηφόρων αηφόρου ανάπτυξης. Χαιρόμαστε διότι η έκθεση αναφέρεται στη συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη αυτών των δικτών, γιατί όπως έχει συζητηθεί, κάποια ζητήματα επιμένουν, Και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όταν νέα δεδομένα προκύπτουν. Πρέπει να έχουμε τα σωστά εργαλεία Τώρα, μας ενδιαφέρει η σωστή ανάλυση να υπάρχει στο δίκτυ για να είμαστε σοφαροί, έτσι ώστε κανείς να μην μείνει στο περιθώριο. Γνωρίζουμε και τις προκλήσεις αυτές που έχουν να κάνουν με το capacity development, το capacity building, να ενισχύσουμε την προσέγγιση μας στο μέλλον για να μπορέσουν οι χώρες να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και πράγματι δεν πρέπει καμία εθνική στατιστική υπηρεσία να, μην, να μείνει πίσω. Θα πρέπει να δούμε και την παροχή των δεδομένων αλλά και τη χρήση αυτών. Είναι εξίσου σημαντικό. και στο μέλλον σίγουρα θα πρέπει να προσαρμόσουμε το πλαίσιο αποτελεσμάτων μας, τον τρόπο με τον οποίο μετρούμε τα αποτελέσματα, έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε στη θέση των χωρών στον κατάλογο των παγκόσμιων δικτών. Ευχαριστώ. thank Να σας υπενθυμίσω ότι το, στο Στρασβούργο υιοθετήσαμε ένα ψήφισμα για την υλοποίηση των ε, στόχων αηφόρου ανάπτυξης όπου στη δεύτερη παράγραφο λέμε ότι καλωσορίζει την έκθεση της υπηρεσίας και της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τους δείκτες για τους στόχους αηφόρου ανάπτυξης, ότι είναι ένα σημαντικό επίτευγμα και καλή βάση για διαπραγματεύσεις. Επομένως βλέπετε ότι η δουλειά αυτή αναγνωρίστηκε από ευρεία πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την έγκριση του ψηφίσματος. Το σημαντικό είναι αυτό το οποίο ε, θέλουμε ως Κοινοβούλιο. Πιέζουμε να υιοθετήσει συνολική προσέγγιση η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γενική Διεύθυνση DEFCO μα είπε ότι θα υπάρχουν εξελίξεις, θα υπάρχει νέα αναπτυξιακή πολιτική για την επίτευξη των στόχων αυτών. Θέλουμε όμως γενικότερα να διαμορφώσουμε την ατζέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα θέματα αυτά. Η Αντιπρόεδρε η κυρία Μογκερίνη, αντιπρόεδρος εξωτερικών σχέσεων και ο κύριος Τίμερμαντς, αντιπρόεδρος εσωτερικών θεμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εργάζονται από κοινού γιατί είναι μια παράλληλη διαδικασία εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής. Ο κύριο Τίμερ μα είπε ότι το θα εγκριθεί η Ατζέντα 2020 έτσι ώστε μέχρι το 2030 να έχουν ενσωματωθεί και οι στόχοι αυτοί. Περιμένουμε λοιπόν ανακοινώσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ατζέντα του 2030. Όλε αυτέ οι στατιστικέ είναι οι σημαντικές. Και όσο περνάει και ο χρόνο, του επόμενου μήνε θα πρέπει να είμαστε σε επαφή εμεί και εσεί για να δούμε τι γίνεται τον Ιούνιο, τον Ιούλιο το... κτλ. Να σα ξαναδώσω το λόγο για να σα πω ότι λαμβάνουμε εκθέσει από τι κυβερνήσει και ξέρετε, κάποιοι είναι καλύτεροι, κάποιοι χειρότεροι, κάποιοι λένε τι πρέπει να γίνει, κάποιοι, κάποιοι κάνουν κρίσιμη αξιολόγηση. Κάποιες εκθέσεις είναι καλύτερες από τις άλλες. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο πρώτος. Με χαρά μου θα μιλήσω πρώτος και θα απαντήσω τις, στις δύσκολες ερωτήσεις τις οποίες είμαι πάντοτε έτοιμος να ακούω. Ευχαριστώ τις ερωτήσεις των κυρίων Ασλάιν και Βίντερ όπως και της Προέδρου στο τέλος και θα απαντήσουμε τη σειρά που έγινε η ερώτηση. Το θέμα της εξισορρόπησης μεταξύ της πολιτικής και του τεχνικού κόσμου. Αυτό είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε στις χώρες μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτή τη δουλειά κάνουμε. Και εδώ το κόλπο ήταν ότι στην ουσία εκ των προτέρων υπήρξε μια συμφωνία για την εντολή πολύ ξεκάθαρη. Η Επιτροπή ε, των Στατιστικών είχε τη δουλειά να εξετάσει τον κάθε στόχο ξεχωριστά, όχι κάτι παραπάνω ούτε κάτι λιγότερο. Κοιτάξαμε λοιπόν τους δείκτες και προσπαθήσαμε να πετύχουμε τους στόχους, όχι να ορίσουμε τους δείκτες. Ήταν πολύ συγκεκριμένη εντολή που ήρθε από όλα τα μέρη του κόσμου, οπότε αυτή η, αυτός ο περιορισμός στην ουσία μας ε, ε, έδωσε τη δυνατότητα να παραμένουμε στο τεχνικό κομμάτι και η απόφαση των επιτροπών, των επιτρόπων τον Μάρτη ήταν κάτι που συμπλήρωσε όλα αυτά ε, και έφτιαξε ένα πακέτο. Έτσι μπορεί κανείς να προχωρήσει είναι ε, το εφαλτήριο αυτό πολύ σημαντικό και θέλουμε να δούμε ε, πόσο επιτυχημένοι θα είναι οι στόχοι για να μπορούμε να τους ε, βελτιώσουμε. Τώρα, το θέμα για την ανάλυση των δεδομένων, την αναλυτική τους παρουσίαση. Θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι όταν σκεφτόμαστε που θέλουμε να επικεντρωθούμε. Η κυρία Μοντέρα μίλησε, πούμε, για την κοινότητα των Ρωμά είναι μια ευαίσθητη κοινότητα και ε, χρειάζονται βασικά στοιχεία για να, τους, για να μετρήσουμε. Ε, δεν μπορεί κανείς να μετρήσει με τους Ρωμά αν δεν έχει στοιχεία για τις γεννήσεις. Ε, χρειάζεται να μπει ένας μηχανισμός σε λειτουργία σε όλες τις χώρες γι' αυτό. Τα κέντρα πληθυσμού επίσης είναι ένα άλλο ζήτημα. Το εξέτασαν το 2010 ε, στην τελευταία συνεδρίαση και έχουμε καλύψει τον περισσότερο κόσμο, όμως σε κάποιες χώρες, όπως η Συρία για παράδειγμα, είναι πολύ δύσκολο να έχουμε οποιαδήποτε μορφή, οποιασδήποτε μορφής συλλογή δεδομένων. Αυτά λοιπόν τα στατικά στοιχεία είναι τα πιο ε, σημαντικά και επιθυμητά στοιχεία που πρέπει να έχουμε για να ξεκινήσουμε. Τώρα, για το πόσο συμμετοχική θα είναι η διαδικασία. Πρώτον, στην συνάντηση, ε, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Στατιστικών είχαμε καμιά διακοσαριά ανθρώπους. Οι περισσότεροι ήταν από ε, ε, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που θέλανε να βοηθήσουν. Υπάρχει σε πολλούς τομείς μεγάλη κινητικότητα για τη μέτρηση. Μπορούμε να υποφεληθούμε από αυτό το ενδιαφέρον. Επίσης υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά της κυβέρνησης. Στην παρουσίασή μου ανέφερα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε τις ε, κυβερνήσει να καταλάβουν ότι η καλύτερη συλλογή δεδομένων, τα καλύτερα δεδομένα οδηγούν και σε καλύτερες αποφάσεις. Θα το καταλάβουν οι κυβερνήσει όταν έχουν τα στατιστικά και θα μπορούν να έχουν τις ε, επιλογές. Ε, αλλιώς δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα. Ελπίζω να απάντησα στις δικέ σα ερωτήσει. Η ερώτηση του κ. νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Είπε ότι ε, πολλά δεδομένα, ε, πολλές χώρες δεν έχουν ε, δηλώσει καθόλου δεδομένα για σημαντικά ζητήματα όπως η ανέχεια. Το πρώτο όπλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο σύγχρονο κόσμο είναι η διαφάνεια. Όταν θα έχουμε μια παγκόσμια έκθεση θα μπορούμε να κάνουμε και τα κατάλληλα ερωτήματα. Είναι δύσκολο τώρα να ψάξουμε. Τα Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει να αποφασίσουν αν πρέπει να κάνουν κάτι παραπάνω, αλλά η διαφάνεια είναι ήδη ένα μεγάλο βήμα. Η δεύτερη ερώτησή σας ήταν λίγο πιο ε, δύσκολη. Πώς διασφαλίζουμε την ακρίβεια και την αλήθεια των δεδομένων. Ε, έχουμε έναν ευρωπαϊκό κώδικα για ηθικής και πρακτικών για τις ε, στατιστικές. Είναι μια πρακτική που μπορούμε να εξάγουμε. Έχουμε επίσης μια διαδικασία εξέτασης και επιθόρηση των συστημάτων στατιστικής πολλών χωρών από άλλους. Υπάρχουν εκθέσεις και πορίσματα που μπορούμε να ε, τα δημοσιεύσουμε. Έχουμε επίση τη διαδικασία για το υπερβολικό έλλειμμα και εκεί υπάρχουν στοιχεία. Υπάρχουν μαθήματα που μάθαμε, ε, που πήραμε μέσα από, την, ε, από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και η Γενική ε, Συνέλευση πριν από δύο χρόνια ενέκρινε τις θεμελιώδεις αρχές ε, για τις στατιστικές που δημιουργήθηκαν στην αρχή στην Ευρώπη, αλλά τώρα είναι αρχές που ασπάζεται όλος ο κόσμος. Αυτά λοιπόν μπορούμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Κοινότητα να τα δώσουμε στον κόσμο. Ε, Αντώνη, η τελευταία ερώτηση για το τι έχει γίνει. Ε, να πω ότι ναι, αυτή ε, ε, η διαδικασία σε αυτό ε, θα οδηγήσει τον Ιούλιο. Αυτό έδειξε η συζήτηση που κάναμε. Τονίσαμε στην ουσία τι ακριβώς χρειάζεται να γίνει. Ωραία, ευχαριστούμε η Μπάρμπαρα. Για να απαντήσω για το εμπόριο, αν περιλαμβάνεται ή όχι στον αντίκτυπο όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και για τις χώρες εταίρους. Καταρχάς να πω ότι το πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνουν όλες οι χώρες είναι τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης να μην τους δουν ως κάτι ξεχωριστό, δηλαδή άλλο αυτό το θεματολόγιο, άλλο η προσφυγική κρίση και ξέρω εγώ, οι εμπορικές συμφωνίες κτλ. η διάσκεψη κορυφής είχε σχεδόν ρεκόρ συμμετοχών. Και αποφάσισαν, μάλλον ήταν πολύ συμμετοχική, με την έννοια ότι σχεδόν όλες οι χώρες συμφώνησαν. Τώρα, η σημασία είναι να είναι συνεπές αυτό, δηλαδή όλοι να εξασφαλίσουμε ότι το αποτέλεσμα στα επόμενα χρόνια θα ε, συμμορφούνται προς το θεματολόγιο αυτών των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό θα είναι αναγκαίο και μπορεί να γίνει με το να αποδείξουμε ότι έχει σημασία, ότι είναι σημαντικό και ότι η προσφυγική κρίση στο εμπόριο είναι συμβατά θέματα. Τι έγινε με παράδειγμα χάρη με τη διάσκεψη για τη Συρία. Δεν μιλάμε για την επίσημη τοξική βοήθεια πια, αλλά και για το πώ μπορεί να αξιοποιηθούν εμπορικέ συμφωνίε για τη διευκόλυνση και τη στήριξη τη διαδικασία, για την συμμετοχή του επιχειρηματικού κλάδου και όλων των άλλων κλάδων. Ουσιαστικά ένα πνεύμα θέλουμε να υλοποιήσουμε, ένα όραμα. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, φυσικά και είναι μια διαδικασία μέσα στην αρχή της μόλις και τα επόμενα 15 χρόνια θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει αλλαγή, πραγματική αλλαγή και σίγουρα το παράδειγμα αυτό είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν. Όλες οι αλλαγές παραδείγματος ε, παίρνουν χρόνο, αλλά είναι εφικτές εάν συμμετέχουν όλοι και αυτό σχετίζεται λίγο και με το ε, ερώτημα της Προέδρου, δηλαδή πώς ε, θα υπάρξει λογοδοσία. Από τη δική μου εμπειρία, για να υπάρξει λογοδοσία, ε, το καλύτερο είναι να έχουμε εθνική λογοδοσία. Δηλαδή, οι κοινωνικοί φορεί, κοινωνικοί παράγοντε, κοινωνικοί των πολιτών, τα κοινοβούλια πρέπει να συμμετέχουν, να μπορούν να χρησιμοποιούν ω αναφορά του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη για τι κυβερνήσει, για του διάφορου φορεί σε σχέση με το πόσο δεσμεύτηκαν, πώς εφάρμοσαν κτλ. Και με πολύ μεγάλη προσοχή επαναλαμβάνουμε ότι αυτοί οι στόχοι δεν είναι των Ηνωμένων Εθνών. Συμμετείχαν και είναι μεγάλη διαφορά η αρχική των κρατών και αυτή τη αποφάσεις. Δεν τους έχουν εφεύρει αυτούς τους στόχους ε, τεχνοκράτες, αλλά είναι αποτέλεσμα, είναι καρπός μακρόχρονων ε, διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών μελών, κοινωνία των πολιτών, ο ιδιωτικός τομέας, ε, πολλοί άλλοι συμμετείχαν. Άρα είναι για το δικό τους το συμφέρον να εφαρμοστεί αυτό το θεματολόγιο και σε οποιαδήποτε ναι εμπορική συμφωνία ή απόφαση περί πολιτικής ε, θα πρέπει να συμμορφώνεται η συμφωνία αυτή με αυτούς τους στόχους και ως προς τον τύπο θα πρέπει να φροντίσουμε και αυτοί να καταλάβουν εγώ έχω εργαστεί κατά το παρελθόν στην Κολομβία και πρέπει να σα πω ότι η συμμετοχή είναι πολύ σημαντική και στι τοπικέ ε, περιφερειακέ εκλογέ. είχαμε εθνικού και τοπικού πολιτικού. που όταν εκλέγονταν δήλωναν με τι θα συμμορφωθούν. Και όταν τέλειωνε η θητεία του αν ήταν στην κυβέρνηση ή αν έπρεπε να επανεκλεγούν, έπρεπε να αποδείξουν τι έκαναν. Και εκεί είναι πολύ μεγάλη σημασία του τύπου μεταξύ άλλων. Είπα ότι θα τα συζητήσουμε στα παγκόσμια βήματα συζήτηση. Ε, ναι, πράγματι, γι' αυτό και είναι σημαντικό. Το πρώτο αυτό φόρουμ θέλουμε ουσιαστικά να αναγνωρίσουμε, αν θέλετε, καταρχά πρωταθλητέ και την προθυμία του, αλλά εντάσσεται και στη διαφάνεια όλο αυτό. Όσοι δεν συμμετάσχουν, ε, μετά θα έχουμε και τη συζήτηση ποιο είναι μέσα και ποιο είναι έξω. Εγώ είμαι αισιόδοξη. Ελπίζω να μην είμαι αφέλη βέβαια. Αλλά ελπίζω ότι όλα αυτά θα οδηγήσουν σε αλλαγές. Και ελπίζω οι Ευρωπαίοι πρωταθλητές να αποδείξουν στον υπόλοιπο κόσμο ότι θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμά μας και τον τρόπο με τον οποίο το κάνουμε. Και θα πρέπει να ακολουθήσουμε τους πρωταθλητές. Και όσοι δεν το έχουν κάνει θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί. Γιατί στη χώρα του ε, δεν έχει μείνει κανεί πίσω, δεν υπάρχει πρόβλημα με την απασχόληση, δεν υπάρχει πρόβλημα με τι διαφορέ μεταξύ των δίφυλων κτλ υπάρχει πολύ ισχυρή συνιστόσα πολιτική υποστήριξης. Δεν θέλουμε να κατονομάσουμε χωρίς δημοσία και να τις ντροπιάσουμε βέβαια, αλλά θέλουμε να έχουμε μια τεχνική συνεργασία μαζί τους για να συμμετέχουν. Σε επίπεδο ΙΕ ε, και τέλο πάντων συνδυασμό ε, αναγνώριση, επονίδηση, ε, συνεργασίας κτλ. ευχαριστώ. Πράγματι, ελπίζω να μας βοηθήσετε και με τη λογοδοσία. θα υπάρξει παρακολούθηση και εμείς θα κάνουμε τη δική μας δουλειά και θα συνεχίσουμε να, να πιέζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει το δικό της μέρη. Σας ευχαριστώ και τους δύο που ήρθατε εδώ. Ελπίζω να παραμείνουμε σε επαφή και να δούμε μέχρι τον Ιούλιο τι γίνεται και να φροντίσουμε να παραμείνει επίκαιρο το θέμα, γιατί αυτό είναι ο κίνδυνος σε δύο-τρία χρόνια να έχει φύγει από τα φώτα της δημοσιότητας. Νομίζω ότι κανονικά όλε οι κυβερνήσει θα έπρεπε να επιθυμούσαν ένα βιώσιμο μέλλον για τη χώρα τους. Και αν μάλιστα το πετύχαιναν, θα ήταν και ιδιαίτερω δημοφιλεί ω κυβερνήσει. Άρα είναι και προ το δικό του συμφέρον. Ευχαριστώ που ήρθατε λοιπόν και οι δύο και θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Λοιπόν, Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό. Θα συνεχίσουμε να το συζητούμε. Πάμε τώρα στο σημείο 8 που είναι η σύναψη της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ από την άλλη αφετέρου. Είναι 6 από τα 15 μέλη της κοινότητας για την ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής, ΚΑΜΑ. Μοζαμβίκη, Μποτσουάνα, Λέσοθο, Ναμίμπια, Νότια Αφρική, Σουαζιλάνδη. Είναι χώρες μεσαίου εισοδήματος. Είναι η πρώτη συζήτηση. Έχουμε γνωμοδότηση ε, που θα εγκρίνουμε εμείς ε, με βάση τη διαδικασία σύμφωνης γνώμης. Φυσικά η ΑΚΕ πηγαίνει στην Αμήμπια σε λίγο καιρό, οπότε φαντάζομαι ότι θα συζητήσουμε περισσότερο για αυτό το θέμα κατόπιν αυτής της ε, συμβολής. Η Νόρμπερτ αντικαθιστά τώρα την ε, εισηγήτρια. Ευχαριστώ, την κυρία Περέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως υπόθηκε ήδη, θα πάμε με την Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή και Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ναμίμπια τον Ιούνιο για να συζητήσουμε και αυτό το θέμα και άλλα. Εκ μέρους ε, του κυρίου Σίλβα Περέιρα, να πω ότι στις 15 ε, Ιουλίου του 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μια συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσεις με έξι από τις ε, ε, χώρες της Μεσημβρινής Αφρικής, η Μποτσουάνα, Λέσοδο, Μοζαμπίκη, Ναμίμπια, Νότια Αφρική και Σουαζιλάνδη ε, χώρες της ε, κοινότητας για την ανάπτυξη της ε, Μεσημβρινής Αφρικής και στο πρώτο κομμάτι του Ιουνίου περιμένουμε την έγκριση αυτής της συμφωνίας. Το Κοινοβούλιο ζήτησε να δοθούν τα συμπεράσματα της ΚΑΜΑ που είναι μία ομάδα από χώρες ε, μεγάλου και μεσαίου εισοδήματος, τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι σημαντικός εμπορικός εταίρος. Αυτές οι χώρες έχουν ένα ενιαίο καθεστώς πρόσβασης 100% duty free πρόσβαση, δηλαδή πρόσβαση χωρίς δασμούς και ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ήδη λοιπόν ε, αυτή την ΣΟΕΣ η οποία θα ε, μπορέσει να θεσπίσει τους όρους ε, για την Συμφωνία Οικονομικής ε, και Εταιρικής Σχέσης. Αυτή η Συμφωνία και Σχέσης. Αυτή η συμφωνία έχει πολλά χαρακτηριστικά. Καταρχάς, έχει μία σύμμετρη που δίνει τη δυνατότητα στους εταίρους από την ΣΟΕΣ να προστατευτούν από τους, ανταγωνιστών. από τους ανταγωνιστές. Οι χώρες ΣΟΕΣ επίσης θα κρατήσουν κάποιο περιθώριο πολιτικής μέσα από δικλείδες ασφαλείας για να προστατέψουν τις εσωτερικές τους αγορές, τον πολιτισμό τους και την τεχνολογία τροφίμων. Τρίτον, ε, έχουμε ε, την κατάργηση των επιδοτήσεων εξαγωγών και δεν υπάρχει απελευθέρωση ε, ε, του ανταγωνισμού ε, που σημαίνει ότι βάσει αυτής της ΣΟΕΣ δεν υπάρχει απελευθέρωση των δασμών. Έτσι είναι πιο εύκολο για τους εξαγωγείς να χρησιμοποιήσουν τα υλικά από άλλες χώρες και μπορεί επίσης σε εξαιρετικές συνθήκες ε, να έχουμε ε, κάποιες, ε, ε δασμούς. Ε, θέλουμε λοιπόν τα μέρη να πληρούν διεθνείς κανόνες και στάνταρτ όπως και περιβαλλοντικούς κανόνες. Η διαδικασία αυτή ε, η συμφωνία αυτή μάλλον ε, θα περάσει μέσα από μια διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των αρχών και των ενδιαφερομένων μερών. Θα ήθελα όμως να σημειώσω ότι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις διαπραγματεύσεις ήταν περιορισμένη και γι' αυτό ενθαρρύνω και παροτρύνω ε, τους ενδιαφερόμενους να πάρουν μέρος στη διαδικασία παρακολούθησης ειδικά. Θέλουμε Βλέπουμε βέβαια με λύπη μας ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένα ένα άρθρο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μιλάμε όμως ε, σε κάποια αναφορά για το δικαίωμα να ληφθούν μέτρα σε περίπτωση παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει αυτές ε, οι ΙΣΟΕΣ να μην χάσουν το σύνδεσμο με την ε, εκνοή της ε, συμφωνίας του Κοτονού το 2020. Επίσης, να πω ότι οι ΣΟΕΣ ήταν, σχεδιάστηκε για να ταιριάζει με το ΣΑΚΟΥ το, την Τελωνιακή Ένωση της Μευθυμπρινής Αφρικής, ειδικότερα για να ενισχύσει το εμπορικό καθεστώς. Θεωρώ ότι οι είναι ε, ένα σημαντικό ε, ε, λιθαράκι για την περαιτέρω ολοκλήρωση αυτής της συνεργασίας για την προώθηση των τεχνικών ικανοτήτων, ας πούμε, για τους κανόνες προέλευσης και τη διευκόλυνση του εμπορίου. Να πάω τώρα σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα εφαρμογής αποτελεσματική εφαρμογή είναι κέρια σημασίας για να μπορέσουμε να πάρουμε τα ωφέλη από την αγορά και τις ευκαιρίες που μας προσφέρει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προβλέψουμε δομές και μηχανισμούς και να τους θεσπίσουμε, όπως επίσης και να διασφαλίσουμε και την διαφάνεια κατά τη λειτουργία τους. Για μένα ίσως πρέπει να παρακολουθείτε με αποτελεσματικό τρόπο σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. αποτελεί αυτό ε, μια επιτακτική ανάγκη. Και επίσης η κατανομή των πόρων είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί θα διευκολύνει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή και την παρακολούθηση. Επίσης θεωρώ ότι θα ήταν ε, καλή ιδέα το Μικτό Συμβούλιο να κάνει εκθέσεις προόδου που θα συζητούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Αφρικανικό Κοινοβούλιο για να αξιολογείται η συμβολή αυτής της εταιρικής σχέσης στο βιώσιμο και δίκαιο εμπόριο, αλλά και στην μείωση της ανέχειας με βιώσιμο τρόπο. Σε αυτό το στάδιο θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρχάς να διασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται για την εφαρμογή αυτής της ε, ε, συμφωνίας. Ποιος είναι λοιπόν ο φάκελος που διατίθεται για την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Επίσης, τι μπορούμε να περιμένουμε από την ε, διαδικασία παρακολούθησης, την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και τη διαφάνεια. Τρίτον, κάποια πρώιμα αποτελέσματα μιας μελέτης που έκανε η ΕΦΠΡΙ ε, δείχνουν ότι αυτή η ΣΟΕΣ θα έχει θετικές αλλά περιορισμένες επιπτώσεις στις ροές του εμπορίου ε, στην αύξηση του ΑΕΠ και τη μείωση της ανέχειας. Μπορείτε να κάνετε κάποιο σχόλιο για αυτά τα αποτελέσματα. Επίσης, ζητούμε από την Επιτροπή να δημοσιεύσει τα τελικά αποτελέσματα ανάλυσης επιπτώσεων ε, αυτής της ΣΟΑΣ ε, πριν εγκριθεί. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους του Πέτρο για την προσοχή σας και να πω ότι μαζί με τους και εισηγητές και όλους τους συναδέλφους αδειμονούμε να δούμε περισσότερα για αυτό το σημαντικό ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σέινφιλντ είναι σκιώδης εισηγητής εκ μέρους του ΕΛΚ. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι παρόν στη σημερινή συνεδρίαση και εκφράζει τη λύπη του γι' αυτό. Επιτρέψτε μου να παρουσιάσω τη θέση του για την έκθεση αυτή. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι η Αφρική είναι μια υπουργός η οποία αναπτύσσεται και κάθε μέρα συστήνονται και διδρύονται νέες εταιρείε. Η οικονομική εταιρική σχέση, η συμφωνία για αυτήν, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο έτσι ώστε να προσεγγίσει η μία ήπειρο στην άλλη όχι μόνο σε ό,τι αφορά στις ανθρωπιστικές πτυχές της σχέσης, αλλά και σε ό,τι αφορά στην οικονομία. Ξέρουμε ότι όλο και μεγαλύτερη πρόσβαση στις αγορές αποκτούν οι χώρες της κοινότητας της νοτιοαφρικανικής ανάπτυξης, SADC. Θα πρέπει όμως να μιλήσουμε για την έλλειψη συμμετρίας στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλάγων. Η συμφωνία περιλαμβάνει πάρα πολλές ασφαλιστικές δικλίδες και μπορούν να τις ενεργοποιήσουν οι χώρες εάν αυξηθούν από οι εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιρετικά γρήγορα και τελικά φανεί ότι διαταράσσουν την ισορροπία στις αγορές. Υπάρχουν κάποιες διατάξεις υπέρ της ανάπτυξη. Για παράδειγμα, έχουμε τους κανόνες προέλευση, οι οποίοι είναι πολύ σαφείς σε ό,τι αφορά τις εξαγωγέ στην κλωστοϊφαντουργία. Και υπάρχουν κάποιες διατάξεις υπέρ της ανάπτυξης, όπως είναι η εξάλληψη των επιδοτήσεων και ενισχύσεων κατά την εξαγωγή. Μεταξύ άλλων. Η ο κλάδος θα διαφοροποιηθεί χάρη στη Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης και θα αυξηθεί και η αξία των προϊόντων. Οι χώρες αυτές, Μποτσουάνα, Λεσότο, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Σουαζιλάνδη, Νότια Αφρική, αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως η έλλειψη μηχανημάτων, η έλλειψη ε, ε, προϊόντων ε, γεωργικών ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση οι δασμοί πρέπει να είναι ευεργετικοί. Και θα πρέπει η συμφωνία να έχει διατάξεις για την βιώσιμη ανάπτυξη και για την ενίσχυση των ανθρωπιστικών προτύπων σε ό,τι αφορά τα εργασιακά και τα περιβαλλοντικά. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η Μαρία Χόιμπουκ και μετά η Λόλα Σάντσεθ. Ευχαριστώ πολύ. Να πω εξ αρχής ε, ότι είχα κάποιες αμφιβολίες και να πω ότι δεν βλέπω κάποιον αυτοματισμό όταν δημιουργούμε ε, τέτοιες συμφωνίες. Δεν υπάρχει αυτοματισμός ε, ότι θα πατάξουμε τη φτώχεια και θα δημιουργήσουμε ανάπτυξη. Η ευρωπαϊκή πολιτική εμπορίου για μένα είναι αμφισβητήσιμη σε αυτό το τομέα. Ε, σε αυτήν εδώ τη Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης με τις χώρες ΚΑΜΑ θεωρώ ότι πήγαμε πάρα πολύ νωρίς σε αμοιβαία απελευθέρωση του εμπορίου. Έχουμε την Κίνα ως πολύ καλό παράδειγμα ε, μιας πολύ καλής οικονομικής ανάπτυξης η οποία προστάτευε πάρα πολύ καιρό την οικονομία της ε, και παρόλα αυτά, παρόλο που είχε ε, ανταγωνιστικότητα μεγάλη και μπορούσε να είναι ανταγωνιστική με καλύτερα ανεπτυγμένες χώρες. Με αυτή λοιπόν την πρώιμη απελευθέρωση θεωρώ ότι η Αφρική θα μπει σε μια δομή που είναι άδικη και δεν θα βοηθήσει στην πάταξη της φτώχειας. Ε, νομίζω ότι υπάρχει πολύ συγκεκριμένος κίνδυνος ως προς την περιφερειακή ολοκλήρωση και δεν συμφωνώ με αυτό που είπε ο εισηγητής ότι προωθείται η περιφερειακή ανάπτυξη. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες θα μπορούσαν να μπουν ε, σε αυτή τη συμφωνία διότι είναι πολλές οι χώρες ε, που συμμετέχουν στην ΚΑΜΑ, είναι 15 οι τρεις καλύπτονται με την Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης για τη Δυτική Αφρική. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά διαφορετικά ε, οικοδομήματα που πρέπει να συνδυάσουμε εδώ και αυτό είναι μεγάλος κίνδυνος, είναι ρίσκο. Ένα άλλο ρίσκο είναι ότι έχουμε λιγότερο ανεπτυγμένε χώρες όπως το Λέσοθο και η Μοζαμβίκη που δεν έχουν κανένα όφελος από αυτή τη συμφωνία ενώ εμείς έχουμε στην Ευρώπη. Επίσης, ε, οι ε, εύκολες χώρες όπως η Μποτσουάνα και η Ναμίμπια ε, με αυτή την οικονομία παίρνουν πολύ καλούς όρους. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα σειράξεων σε αυτή την ίδια την περιοχή. Ένα άλλο θέμα για μένα είναι ότι αυτή η οικονομική η ε, συμφωνία δεν δίνει κάποιο κίνητρο για διαφοροποίηση να ε, έχουμε άλλα προϊόντα. Έχουμε όλο και πιο πολύ ε, τα ψάρια. Επίσης έχουμε τα στάνταρ της Ευρώπης για την υγιεινή, για το περιβάλλον πράγματα που υπάρχουν στην Ευρώπη. Η δημιουργία αξία θα γίνει δηλαδή στην Ευρώπη και όχι επιτόπου στις χώρες αυτές που χρειάζονται κάτι τέτοιο άμεσα ε, σε επίπεδο ας πούμε εμπορίου πρώτων υλών. Και αυτό είναι ένας από τους μεγάλους κινδύνους της βιομηχανοποίησης. Επίσης, ε, ε, αυτό το είδαμε και στη δεκαετία του 80 και του 90. Ένα άλλο θέμα είναι η διανοητική ιδιοκτησία. Ε, η Αφρικανική Ένωση εργάζεται επ' αυτού και φαντάζομαι ότι με αυτή τη συμφωνία ε, θα, έχουν, θα έχει περιοριστεί το πεδίο χειρισμών που έχουν. Επίσης, οι για το περιβάλλον θεωρώ ότι και εδώ Υπάρχει ε, πιθανότητα να έχουμε προβλήματα, διότι ε, όταν υποσχόμαστε κάτι θα πρέπει να το δίνουμε τελικά. Ας πούμε, ε, ε χρειαζόμαστε πολύ συγκεκριμένους νομικά δεσμευτικούς κανόνες. Ε, σήμερα το, πρωί, το απόγευμα μιλήσαμε για την βιομηχανία ένδυσης. Θέλουμε στο εργασιακό επίπεδο λοιπόν τέτοιους κανόνες και θα πρέπει να επαναληφθεί και εδώ. Επίσης, Υπάρχει και ένα άλλο αμφισβητούμενο σημείο ε, κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα ε, χειρισμών ε, που να, αφήν, να αφήνουν το περιθώριο δηλαδή για χειρισμούς σε αυτές τις χώρες που χρειάζονται άμεσα τα χρήματα αυτά. Η κοινωνία των πολιτών επίσης είναι κάτι για το οποίο συμφω... με το οποίο συμφωνώ με τον συνάδελφο που αναφέρθηκε πάρα πολύ στο θέμα αυτό. Επίσης, τα ντόπια κοινοβούλια δεν ενεπλάκησαν πολύ και επίσης για φορολογικά θέματα σε αυτή τη συμφωνία γίνεται πολύ ε, σύντομη αναφορά. Πολλές νοτιοαφρικανικές ε, χώρες ε, έχουν πάρα πολύ σημαντικό ε, τομέα γεωργίας και αυτός είναι το φορολογικό ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς. Ε, θέλουμε διαφανείς κανόνες και στάνταρτ αναχώρα και καταγραφή αναχώρα. Αυτά είχα να σχόλια και κριτική και περιμένουμε και τις τροπολογίες για να τα καταθέσουμε πιο συγκεκριμένα. Thank you, Lola Ευχαριστώ πολύ, Λίντα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η συμφωνία αναπαράγει την νεοαπικιοκρατική λογική η οποία δίνει πρωτοκαθεδρία στην εταιρεία του Βορρά σε βάρος την ευημερία, της ευημερίας του κόσμου του Νότου. Και αφιβάλλουμε για τον τρόπο με τον οποίο έγινε αντικείμενο διαπραγμάτευσης η συμφωνία. Δεν μπόρεσε η κοινωνία των χώρων του Νότου να συμμετάσχει ούτε να ζητηθεί η γνώμη της, όπως ήθιστε. Πολύ μας ανησυχεί το, ο αρνητικός αντίκτυπος που θα έχει ε, στη ροή παράνομων κεφαλαίων και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πριν από λίγους μήνες, στην Επιτροπή ΙΝΤΑ αυτού του Κοινοβουλίου παρουσιάστηκε μια έκθεση για τη σχέση μεταξύ των εμπορικών σχέσεων ε, τέτοιου τύπου και συμφωνιών με τη φορολογική απάτη και το ξέπλυμα χρήματος. Και η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η απελευθέρωση του εμπορίου υπηρεσιών και προϊόντων με τις αναπτυσσόμενες χώρες αυξάνει την απειλή ξεπλήματος χρήματος και ε, αυξάνει το κίνδυνο να υπάρξει ροή κεφαλαίων παρανόμης προέλευσης από τις αναπτυσσόμενες χώρες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί ιδιαιτέρως και ειδικότερα στην πολιτική ομάδα, η οποία ανησυχεί ιδιαιτέρως για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις αναπτυσσόμενες χώρες και δεν θεωρούμε ότι ε, αυτή αυτές οι συμφωνίες δίνουν λύσεις. Αντιθέτως, οξύνουν τα προβλήματα γιατί οδηγούν στην, στον προσπορισμό των γεών και των εδαφών από διάφορες πολυεθνικές ε, με διάφορα προσχήματα. Και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όλο αυτό το ζήτημα της ε, καταστρατήγησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για όλους αυτούς τους λόγους η ομάδα μου θα είναι κατά της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης. Το εμπόριο πράγματι είναι εργαλείο για την ανάπτυξη, αλλά όχι όποιο εμπόριο και να είναι. Πόσο μάλλον όταν το εμπόριο το μόνο που κάνει είναι να υπηρετεί την νεοφιλελεύθερη λογική που ε, επιβαρύνει το περιβάλλον, επιβαρύνει τα δικαιώματα των κοινωνιών και ε, επωφελεί μόνο τους μεγάλους ομίλους. Ευχαριστώ. Äh Κύριε Ζέλερ, ευχαριστώ συνάδελφοι. Εδώ ακούμε πολλή ιδεολογία και στις θέσεις και στη γνωμοδότηση θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Ε, το ε, θέμα είναι ότι όλοι έχουμε τεθεί ενώπιον αυτής της συμφωνίας. Πρόσφατα ήμασταν σε μια περιφερειακή διάσκεψη ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΚΕ στη Νότια Αφρική και εκεί έπαιξε αυτό το θέμα της δημιουργίας της σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΣΟΕ. Έπαιξε σημαντικό ρόλο. Να πω λοιπόν ότι ε, η βάση που έχουμε ως τώρα η συμβατική με τα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού ε, θα εκπνεύσει το 2020. Και υπάρχουν κάποιες διαπραγματεύσεις ε, που έχουν ξεκινήσει για την επέκτασή της, αλλά υπάρχουν πολλές αμφιβολίες κατά πόσο θα καταλήξουμε σε μια σύμβαση. Στο πλαίσιο λοιπόν και υπό την αιγύδα της Συμφωνίας ε, Κοτονού οι χώρες ε, ΑΚΕ, Αφρική, Καραϊβική και Ειρηνικού ε, πάρα πολλούς στόχους συνδυάζουν πράγματα που έχουμε συμφωνήσει με τη Συμφωνία Κοτονού για την οικονομία, για το εμπόριο. Όλα αυτά θέλουμε ε, μαζί με τη συνεργασία να τα αποτυπώσουμε με μία ε, σύμβαση, μία συμφωνία. Τώρα το ότι έχουμε ε, αυτή τη συμφωνία και με χώρες της Αφρικής, νότιας, ανατολικής, και ε, δυτική είναι πολύ σημαντικό. Στη Μεσημβρινή Αφρική υπάρχουν 15 ε, κράτη και σε αυτή τη συμφωνία συμμετέχουν τα 6. Ε, μόνο τα 6 ζήτησαν να υπάρχει κάποια συμβατική σχέση. Δεν ξέρω κατά πόσο η κοινωνία των πολιτών αρκεί, η συμμετοχή που είχε δηλαδή, για να μπορέσουμε να θεωρήσουμε ότι είναι υπεύθυνη η στάση τους ε, ως προς αυτή τη σύμβαση. Ε, επίσης, έχουμε την τελευταία απολυταρχική ε, μοναρχία σε μία από τις χώρες αυτές. Ε, δεν υπάρχει κοινοβούλιο, μόνο ο βασιλιάς αποφασίζει, άρα... Ήταν δύσκολο κάποιες φορές να έχουμε κοινοβουλευτικές δομές, ειδικά εφόσον έχουμε τις πιο φτωχές χώρες Στη Σουαζιλάνδη συγκεκριμένα ε, ε, υπήρξε αυτό το πρόβλημα με τη μοναρχία. Ε, είναι σημαντικό λοιπόν επίσης να θέσουμε το θέμα της ενέργειας, ας πούμε στη Σουαζιλάνδη και σε πολλές από αυτές τις χώρες έχουμε μια περιφερειακή συνεργασία η οποία ζητήθηκε μεν, αλλά δεν υπάρχει λογική βάση, γιατί είναι πολύ επιφανειακή αυτή η περιφερειακή συνεργασία, δεν ε, έχει δημιουργηθεί και περιορίζεται σε διμερείς ε, συμβάσεις και συμφωνίες. Άρα ε, θα έπρεπε να γίνει περιττέρω διαπραγμάτευση για κάτι τέτοιο. Επίσης, η η Σουαζιλάνδη έχει από το, μέχρι το 2024 μια σύμβαση ε, με την Νότια Αφρική για παράδοση ενέργειας, όμως η Νότια Αφρική δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα επεκταθεί αυτή η συμφωνία και θέλουν να φτιάξουν ε, μεταλλεία για ε, άνθρακα γιατί χρειάζονται τις πρώτες ύλες και επίσης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητήθηκε το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες όμως τελικά είναι πολύ ακριβές. Αυτό ήταν το πλαίσιο μέσα στο οποίο έπρεπε να συζητήσουμε με αυτές τις χώρες εταίρους και γι' αυτό για αυτά τα θέματα χρειαζόμαστε μια συμβατική βάση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτοί οι ΣΟΕΣ ε, ε, ε, με την κάμα που έχουμε συζητήσει εκεί με τα διάφορα φορά, αν τελικά εδώ κριθεί αρνητικά, θα, είναι δύσκολο να προχωρήσουμε γιατί είμαστε ο μοναδικός θεσμός που μπορέσαμε να έχουμε και συντονίσει μια σχέση μεταξύ αυτών των 15 ε, χωρών. Σταματήστε λίγο γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα με την αγγλική. Συγγνώμη, μισό λεπτό, υπάρχει πρόβλημα με την αγγλική μετάφραση. Όχι, δικό μου ήταν το πρόβλημα, λέει η πρόεδρος. Συνεχίστε. Θα είχαν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση την ευθεντία της και την εξουσία της, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, το κύρος της μάλλον. Ε, και θα μέναμε με τις διμερείς σχέσεις που ήδη υπάρχουν. Αυτά είναι ε, τα προβλήματα και οι κίνδυνοι που ήδη έχουν αναφερθεί. Ας πούμε το θέμα της Ζάμπια που ανήκει σε αυτή την ε, κοινότητα για την ανάπτυξή της Μεσηβρινής Αφρικής. Εκεί ε, οι πρώτες ύλες ε, ας πούμε από κινέζικες εταιρείες και υπάρχει ε, πάρα πολύ μεγάλο παράνομη δράση εκεί και με αυτές τις διαδικασίες θα μπορούσαμε τουλάχιστον να επηρεάσουμε τέτοιες καταστάσεις. Κάτι που δεν θα μπορούσαμε αλλιώς. Ε, νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να υπερψηφίσουμε γιατί ε, θα μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να βελτιώσουμε τα πράγματα και χρειάζεται βελτίωση και έτσι θα γίνει, αλλά δεν θα πρέπει εκ των προτέρων να θεωρούμε ότι έχουν καταρρεύσει ε, όλες οι πιθανότητες που έχουμε να έχουμε περισσότερη επιρροή σε αυτή την περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν πολλά ζητήματα ε, και ερωτήσεις προς τις ε, δύο γενικές διευθύνσεις ε, DEFCO και TRADE. Πρώτα η εκπρόσωπος της ΓΔ TRADE. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για τη χρηματοδότηση η Ρένα θα τα πει, γιατί είναι ειδικότητά της να δώσω λίγες απαντήσεις που ελπίζω ότι θα καλύψουν τα βασικά. τα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση σήμερα. Αλλά πρώτα κάποια τεχνικά. Κάτι το οποίο πάρα πολύ εύγλωτα είπε ο κύριος Νόιζερ. Τεχνική ασυμμετρία θα τη χαρακτήριζα. Να τονίσω ότι πρόκειται για μια συμφωνία που έχει έξι ασφαλιστικές δικλείδες που κινητοποιούνται και ενεργοποιούνται πάρα πολύ εύκολα, το τονίζω αυτό. Εύκολα λοιπόν ενεργοποιούνται σε όλες τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέση. Έχουμε έξι αυτή τη φορά γιατί θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ε, Λεσότο, η Αφρική, τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, παλιότερες και τις υπόλοιπες. Άρα θα ενεργοποιούνται με λίγη προσπάθεια, αρκεί να υπάρχει μια απειλή για ασφαλιστικές αυτές δικλείδες ε, δεν είναι, αν θέλετε, ασφαλιστική δικλία τύπου ΠΟΕ. Τώρα για τους κανόνες προέλευσης κάποιος μίλησε. Να σας πω ότι όταν έφυγε η Αγγόλα, εμείς ήμασταν ε, η βάση και ιδίως για το Λεσότο. Ε, άρα η γλωσσεφαντουργία είναι ένας τομέας που θέλουμε να έχουμε εξαγωγή, αν θέλετε, προστέμενη αξία. Και δεν μιλώ μόνο για τα υφάσματα. Η συμφωνία στόχο έχει την προστέμενη αξία. Γιατί θα δείτε ότι σε σχέση με το τι κάνουν καλύτερα και μιλάω για το γεωργικό σκέλο, σε σχέση με το γεωργικό σκέλο, ο φίλε, η περαιτέρω απελευθέρωση σε σχέση με το τι υπήρχε για του δικού του σκοπού για όλου τον κόσμο, δηλαδή ήταν μόνο 2% να το έχετε υπόψη αυτό το ποσοστό. Ε, πολύ ευαίσθητο το θέμα της γεωργίας. 65 με 70% του πληθυσμού ζει από τη γεωργία σε αυτές τις χώρες. Άκουσα πολύ προσεκτικά τις δηλώσεις που υπερβαίνουν βέβαια τις τεχνικές πτυχές και μία από αυτές τις πτυχές είναι περιφερειακός χαρακτήρας. Εναρμόνιση, σάκο. Θέλουμε να προσιλητήσουμε, θέλετε να τραβήξουμε κοντά μας μια μεγάλη χώρα όπως είναι η Νότια Αφρική. Δεν θέλουμε να παραμείνουμε στι ε, παλιού τύπου συμφωνίες, εμπορικέ συμφωνίε. Λοιπόν, θέλουμε μια συμφωνία υπέρ της ανάπτυξης με την Νότια Αφρική, με ένα Μίμπια, Μποτσουάνα, τι χώρες περιοχής, ε, άρα πιέσουμε στα τα πάνω τις χώρες μεσοσοδήματος, όπως είναι και η Σουαζολάντ, 10.000 ε, κατά κεφαλήν εισόδημα. Και εδώ έρχομαι σε αυτό που εκφράσατε και που πρέπει και εμείς να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Δηλαδή την ανάγκη να έχουμε καλή παρακολούθηση, καλό έλεγχο. Η συμφωνία θα κριθεί από την εφαρμογή τη και από την υλοποίηση της εφαρμογή τη. Πρέπει να σας πω ότι άκουσα πολύ ξεκάθαρα την ανάγκη συμμετοχή κοινωνικών των πολιτών. Ναι, δυστυχώ! δεν συμμετείχε τόσο πολύ στι διαπραγματεύσει κοινωνικών πολιτών. Αν είμαστε αξιόπιστος εταίροι, τόσο που κάνουμε ό,τι μπορούσαμε και στις διάφορες ομάδες εργασίας για να συμπεριλάβουμε αυτό το οποίο εγώ θα έλεγα κοινωνία των πολιτών. Και η πραγματική κοινωνία των πολιτών πρέπει να συμμετέχει στην παρακολούθηση. Και πρέπει να μας βοηθήσετε και εσείς στο Κοινοβούλιο, διότι υπάρχει περιορισμένη εξοπιστία. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε περισσότερο στους διαπραγματευτές από ό,τι μπορούμε να επηρεάσουμε. Είναι σημαντικά τα μηνύματα που δίνουμε Άρα θα μπορούσαμε στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα, όπως φορολογία, πολύ σημαντικό ζήτημα. Αλλά ξέρετε, αυτή η συμφωνία έχει περιορισμένο παιδί εφαρμογή. Γιατί θέλαμε να εστιάσουμε στον αναπτυξιακό πυλώνα και στον πυλώνα των αγαθών. Για το πρωτόκολλο γεωγραφική ένδειξη. Δεν υπάρχει IPR, δηλαδή πνευματική διοκτησία, ανταγωνισμό ε, κτλ. Το πρωτόκολλο για τη γεωγραφική ένδειξη μόνο με την Νότια Αφρική έχει υπογραφεί, που είναι ο μόνο εταίρο. Θέλουν τι γεωγραφικέ ενδείξει. Και αυτό είναι τεράστιο μήνυμα και προ τη ΣΥΠΑ και για το θεματολόγιο του ΠΟΕ. Και μα ικανοποιεί ιδιαίτερα αυτή η εξέλιξη. Τώρα, είπα, δίνουμε σημάδια, μηνύματα εκπέμπουμε. Τι μήνυμα θα στείλουμε σε αυτή την περιοχή και σε αυτές τις χώρες. Ότι η Ευρώπη προχωρά και λέει ναι, Θέλουμε να συμφωνήσουμε μαζί σας, να περάσουμε σε αυτή τη συμφωνία. Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα. Γιατί προσπαθούν αυτές οι χώρες. Ίσως να μην είναι αυτή η συμφωνία πανάκια για όλα τα προβλήματα, αλλά προσπαθούν να βγουν από το μονομερές αυτό καθεστώς, να έχουν κάτι διαφορετικό, να έχουν κάτι που, πώς να το πω, είναι μια ευρεία αναπτυξιακή συμφωνία, αλλά συμφωνία. Να μην τους απογοητεύσουμε λοιπόν. Πιστεύω ότι οι συζητήσεις που θα έχετε στην Αμίμπια θα σας δείξουν πόσο έντονες είναι ε, οι απόψεις τους για αυτή τη συμφωνία, η οποία ήρθε μετά από μια μακρά περίοδο που είχαμε, αν θέλετε, μία συζήτηση μία κουόντων, σε ότα μία κουόντων οι υπηρεσίε δεν ήταν στο πέντε εφαρμογή και πολλά άλλα πράγματα που θέλαν όλοι, αλλά παραδείγματο χάρη δασμολόγητα, προϊόντα κτλ. Ε, μπορώ να σα δώσω στοιχεία, αλλά δεν θα βοηθήσουν. Μόνο ε, αρκεί να ακούσετε για τα σπεριδοειδή να σα μιλάει ένα Νοτιοαφρικανό και ότι τα πορτο, οι πορτοκαλάδες που πίνετε στην πλειοψηφία τους προέρχονται από τη Νότια Αφρική τα πορτοκάλια και δεν θέλουν αδασμολόγητα ε, προϊόντα. Λοιπόν, ε, υπάρχουν πολλά άλλα θέματα που δεν πρέπει να τους πούμε. Σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Ε, φύγετε. Αντίθετα, θέλουμε να ανοίξουμε τις αγκάλες μας και να τους πούμε, ελάτε. Είναι δύσκολο, αλλά θέλουμε να πετύχουμε μια καλή συμφωνία, αλλά μόνο μαζί θα την πετύχουμε. Δεν μπορούμε να τους την εξαγάγουμε και να τους πούμε τώρα, ορίστε, την εφαρμόζετε. Επίσης, και τα άλλα που είπατε είναι πολύ σημαντικά. Να δώσω τώρα το λόγο στην Ιρένη. Thank you, Sandra. Thank you, Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, καλά, καλησπέρα σε όλους. Πάντοτε είναι δύσκολο το εγχείρημα να μιλάω μετά τη Σάντρα, γιατί πείθει εξαιρετικά καλά. Θα προσπαθήσω όμως κάποια θέματα να τα θέσω. Σας ευχαριστώ που ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών. Είναι σημαντικό κομμάτι αυτής της συμφωνίας. Υπάρχει ένα κεφάλαιο με το οποίο δεσμεύουμε τις δύο, τα δύο μέρη. Δεσμεύονται τα μέρη να συνεργαστούν και να στηρίξουν διάφορους κλάδους, πολλούς και επικύλους και εκτεταμένους. Φαίνεται αυτό στην συμφωνία. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δεσμευμένες να στηρίξουν τις χώρες που αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην εφαρμογή και την υλοποίηση όλων αυτών. Και όλα αυτά θα γίνουν βάσει των διαδικασιών ε, και των κανόνων και κανονισμών και διατάξεων και φυστάμενων εργαλείων που διέπουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τον προπολογισμό μας. Μεταξύ άλλων και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο βέβαια θα πρέπει να στηρίξουμε τις μεταρρυθμίσεις που ετοιμάζουν οι χώρες αυτές για να μπορούν να εφαρμόσουν το ΙΠΑΣ. Και έχουμε ξεκινήσει τις συζητήσεις με τις κυβερνήσεις, μέσω των αντιπροσωπιών μας στις διάφορες χώρες, για το πώς θα έχουμε εξατομικευμένη στήριξη ανά χώρα. Aid for Trade, ο ορισμός αυτό από τον ΩΣΑ είναι πολύ σημαντικός. Τεχνική βοήθεια για εμπορική πολιτική, κανονισμούς, για υποδομές σε σχέση με το εμπόριο, για τη δυνατότητα χτισήματος δεξιοτήτων, για τις προσαρμογές ε, που σχετίζονται με το εμπόριο και οποιαδήποτε σε άλλες πτυχές της συνεργασίας που ε, υπάρχει μεταξύ των μερών και είναι ενταγμένη ε, στην αναπτυξιακή στρατηγική. Αυτή είναι η βάση του διαλόγου με τις κυβερνήσεις. Τα εργαλεία που έχουμε εντοπίσει είναι τα εθνικά ενδεικτικά προγράμματα, το 11 BTF, agribusiness, στήριξη στις γεωργικές επιχειρήσεις, στάνταρτ και κανόνες και πρότυπα για τις υποδομές μεταξύ άλλων Έχουμε και τα σχέδια υλοποίηση και εφαρμογή, που είναι μια ανάλυση των συγκεκριμένων αναγκών σε εθνικό επίπεδο. Ανάγκες που θα προκύψουν από την εφαρμογή. Προσπαθούμε να προβλέψουμε τις ανάγκες, να στηρίξουμε τα σωστά μέτρα στη σωστή χώρα και έχουμε και το περιφερειακό πρόγραμμα δικτών για τον Ινδικό ωκεανό και την, ε, Δυτική, και την Ανατολική Αφρική και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό οι, χώρες ξεχωριστά. Ένα σωρό προγράμματα έχουμε που ε, υλοποιούνται και που εξελίσσονται. Έχουμε και το ε, πρόγραμμα διευκόλυσης του εμπορίου. Κάθε χώρα μπορεί να προτείνει μια, ένα συγκεκριμένο θεματολόγιο μια ατζέντα για την ολοκλήρωση του εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να έχει και η κονδύλια από το περιφερειακό πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε πάνω σε μια πρόταση της Ναμίμπιας. Να σας μιλήσω πιο συγκεκριμένα. Ε, εθνική η μόνο απευθυντική θηρίδα στην Αμήμπια για, την, ε, για τον εξυγχρονισμό της βιομηχανίας. Στο Λεζότο μιλούμε για τα στάνταρ ποιότητας, για να υπάρχει ένα κέντρο στο οποίο μπορούν να απευθύνονται οι επιχειρήσεις. Όλες αυτές, όλα αυτά είναι μικρά παραδείγματα μέσα σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα που αναπτύσσει κάθε κυβέρνηση. Θα είμαι βέβαια στη διάθεσή σας για ερωτήσεις, αλλά θα ήθελα να πω ότι στηρίζουμε και τη ΣΑΝΤΕΚ ως περιφερειακή οργάνωση και θέλουμε να εφαρμοστεί και να ελοπιθεί το πρωτόκολλο το σχετικό. Έχουμε χρηματοδότηση 90 εκατομμύρια ευρώ για την περιοχή και έχουμε 600 εκατομμύρια ευρώ που θα ε, αναμειχθούν και με εθνικά κονδύλια και με ίδιους πόρους για εθνικά έργα υποδομής μεταξύ άλλων σε όλες τις χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Αφρικής ευρύτερα. Μας ενδιαφέρει να στοχεύουμε τους σωστούς τομείς που έχουν περισσότερες δυνατότητες να οδηγήσουν σε εξαγωγές από τις χώρες αυτές προς την Ευρώπη. Και δύο λόγια να πω για την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών από πλευράς μας. Κατά την κατάρτιση οποιοδήποτε προγράμματος έχουμε ένα σύστημα τακτής διαβούλευσης με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Το κάνουν οι αντιπροσωπείες μας αυτό σε κάθε ενδιαφερόμενη χώρα. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ. Νόρμπερτ, θέλεις να σχολιάσεις, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Να κάνω μια σειρά παρατηρήσεις για τη συζήτηση και να ευχαριστήσω και την Επιτροπή για την ξεκάθαρη θέση της, διότι έχει τονίσει κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Όντως, η κοινωνία των πολιτών πολύ λίγο ε, ε, ενεπλάκη και όντως λίγο ασχοληθήκαμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με αυτή την ε, ε, συμφωνία Εμπορίου δύσκολα θα αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια. Όλα αυτά ισχύουν, όμως υπάρχουν και κάποιες δυνατότητες που και στο παρελθόν δεν χρησιμοποιήθηκαν αρκετά όπως ε, η Συμφωνία Κοτονού, όπου τα δικαιώματα τα ανθρώπινα λίγο αναφερόταν, όμως ε, κατά την εφαρμογή και την παρακολούθηση χρησιμοποιήθηκαν δυνατότητες δεν έχουμε τον κίνδυνο να έχουμε νεοαπικιακές δόμες. Ε, πώς θα αντιμετωπίσουμε χώρες οι οποίες είναι δημοκρατικά δομημένες, αλλά που δεν είναι ε, δημοκρατικά δομημένες. Ε, εμείς, αν θέλουμε ως Ευρωπαίοι να δούμε τι έχουμε διαπραγματευτεί μεταξύ μων και αυτών, αν είμαστε ειλικρινείς, θα ε, παραδεχτούμε ότι λίγα πράγματα, πολύ λίγα πράγματα ε, υπάρχουν ας πούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως είναι και οι κυβερνητικέ οργανώσεις όμως πέρα από όλες τις κόκκινες γραμμές που τραβάμε ε, σε όλες τις συμφωνίες εμπορίου και δικαίως θα πρέπει να σκεφτούμε με ποιο τελικά θα πρέπει να διαπραγματευτούμε και θα έχουμε να διαπραγματευτούμε, θα πρέπει να έχουμε και πράσινες γραμμές οι οποίες ε, θα μας βοηθήσουν και με θετικό τρόπο. Αλλιώς ε, δεν θα μπορούμε να έχουμε περισσότερα ε, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, την Βραζιλία, την Ινδία. Αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να τα θέσουμε σε συζήτηση. υπήρξε μια έντονη συζήτηση μεταξύ του Πέτρο και των Σκιωδών ε, και νομίζω ότι ε, δικαίωση έγινε αυτό γιατί πρέπει εντατικά να ασχοληθούμε με αυτή την παραδειγματική συμφωνία. Ευχαριστούμε. Θα συζητήσουμε την έκθεση στην επόμενη συνεδρίασή μας τον Ιούνιο και θα υπάρξει και το σχέδιο γνωμοδότησης από τον ε, εισηγητή για τη γνωμοδότηση. Τώρα, συνάδελφοι, έχουμε ένα πρόβλημα. Υπάρχει το σημείο 9 για τον προϋπολογισμό. Περιμέναμε τον εισηγητή, τον κύριο Γκάιερ, όμως έχει κολλήσει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και δεν θα μπορέσει να έρθει σήμερα. Ο κύριος Ντέβα επίσης, ο εισηγητής μας δεν είναι εδώ. Ζήτησε την κυρία Ραντήλ να τον, κυρία να τον αντικαταστήσει. Όμως δυστυχώς κυρία Ραντήλ φαίνεται ότι θα πρέπει να αναβάλουμε το σημείο αυτό μέχρι τον Ιούνιο και δεν, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε τον κύριο Γκάιερ 45 λεπτά μέχρι να έρθει. Λυπάμαι λοιπόν, ε, πρέπει να ακυρώσουμε, να αναβάλουμε μάλλον αυτό το σημείο της μερίσας διάταξης μέχρι τον Ιούνιο. Ήδη το θέμα της Σομαλίας έχει ακυρωθεί, άρα λίγη κάπως πρόωρα η συνεδρίασή μας σήμερα και αύριο το πρωί στις 9 θα ξαναβρεθούμε εδώ για τις ψηφοφορίες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τους ε, διερμηνείς. Όλοι θα πάμε σπίτι λίγο νωρίτερα από ό,τι σχεδιάζαμε.